λοιπόν και ελπίζω στο μέλλον να είστε τόσο οργανωτικός όσο ήσασταν και σήμερα. Ε, ε, Σας ευχαριστώ κυρία μου. Εύχομαι και εγώ η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραμείνει το ίδιο αγαστή όπως απόψε. Ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας. Υπάρχει μία πρόταση ψηφίσματος για το θέμα αυτό και εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος αυτού. Η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο. Ευχαριστώ όλες και όλους και σας εύχομαι καληνύχτα. Η επόμενη συνεδρίαση αρχίζει αύριο 17 Ιουνίου, 5η στις 9 το πρωί μέχρι τις 13 και το απόγευμα